Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 13 μετά το μεσημέρι και από τις 15 έως τις 17 με την ημερήσια διάταξη